Liebe Kolleginnen und Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλοχαιρετήσω και σας καλωσορίζω στη σημερινή μας συνεδρίαση. Πρωτού περάσουμε στην ημερήσια διάταξη, θα ήθελα στον συνάδελφό μας Ότμαρ Κάρας, που τον είδα να μπαίνει στην αίθουσα μόλις πριν από λίγο, να τον συγχαρώ για το ότι ανέκτησε την υγεία του όπως ελπίζω και ανέρωσε πλήρως. Ξέρουμε ότι είχε κάποιες ε, πολύ δύσκολες εβδομάδες ε, που πέρασε και χωρίς να φταίει τίποτα. Αλλά αυτό συμβαίνει στη ζωή. Όταν πλήττεται κάποιος όταν τον χτυπάει η ατυχία είναι σοβαρό το συμβάν. Και τώρα, ακριβώς τώρα που περνάμε στην αποφασιστική τελική φάση και που μπορούμε να βασιστούμε στην ε, συνεργασία σου, έχει διανεμηθεί η ημερήσια διάταξη, δεν υπάρχουν κάποιες άλλες αλλαγές ή επιθυμίες. Έχουμε πλήρη διερμηνία. Σας έχουν διανεμηθεί επίσης και τα πρακτικά των συνεδριάσεών μας στις 28 Φεβρουαρίου, 3ης και 14ης Μαρτίου και εδώ δεν υπήρξαν αλλαγές ώστε πάλι μπορούμε αμέσως να περάσουμε στην πραγματική συζήτηση της ε, τελικής έκθεσης της Περβάνς Μπερέσα. Ως πρόεδρος δεν έχω κάποιες ανακοινώσεις να κάνω. Ίσως θα ήθελα όμως για εκείνους που δεν ήταν παρόντες να πω σύντομα δύο λόγια για τη χθεσινή συνεδρίαση. Είχαμε τη χαρά και την τιμή ταυτόχρονα να έχουμε τον Φιλ Αγγελίδης ανάμεσά μας εχθές. Ο Φιλ Αγγελίδης είναι πρόεδρος της Financial Crisis Inquiry Commission της Διακριβωτικής Επιτροπής για την Χρηματοοικονομική Κρίση που θεσπίστηκε, συγκροτήθηκε στη ΣΥΠΑ το 2009 και στις αρχές Φεβρουαρίου φέτος υπέβαλε την τελική της έκθεση. Η τελική έκθεση είναι ένα πολύ διεξοδικό εκτενές έγγραφο πάνω από 500 σελίδες. Από τότε που δημοσιεύθηκε, δημοσιοποιήθηκε είναι στον κατάλογο των ευπόλυτων, των best sellers στη ΣΥΠΑ. Μας παρουσίασε τα συμπεράσματα και τις αναλύσεις του ο Φίλ Αγγελίδης. Η στοχοθέτηση αυτή τη Επιτροπή ήταν διαφορετική από τη δική μα. Μόνο με τα αίτια τη κρίση έπρεπε να ασχοληθούν. Να, δεν χρειαζόταν να δώσουν πολιτικέ συστάσει ε, από τα συμπεράσματά του. Παρότι, συμπεράσματά τους, παρότι έμεσα φυσικά η συζήτηση για αυτά τα θέματα για ε, την οποία ο Φιλ είχε συμμετάσχει δείχνει την ανάγκη αυτών. Τώρα, Είχα ε, υποθέσει και είχα πει ότι πολύ εξειδικευμένα και ε, ανοιχτά η Επιτροπή μας ε, θα συζητούσε αυτά τα θέματα όπως και το έκανε και πλούσιο υλικό είχαμε στα χέρια μας. Μέχρι σήμερα η Wall Street, το αμερικανικό χρηματιστήριο, μεγάλο αριθμό νομικών ομομαθών απασχόλησε για να βρουν κενά σε αυτή την έκθεση. Δεν μπόρεσαν ούτε ένα κενό να βρουν σε αυτή την έκθεση όμως ώστε μπορεί κανείς να υποθέσει και να πει ότι πραγματικά τα στελέχη αυτής της Επιτροπής, 90 μέλη, συνεργάτες και μέλη, εργάστηκαν πολύ αποτελεσματικά και σε βάθος. Σας συνιστούμε την ανάγνωση. Μπορεί κανείς να αποκτήσει και το βιβλίο, κοστίζει 13,99 ευρώ. Νομίζω καθένας μπορεί να το αγοράσει, είναι προσιτή τιμή. Και τώρα περνάω στο ουσιαστικό θέμα της σημερινή μας συνεδρίασης της σημερινής μας συνεδρίασης. Ευθύ εξ αρχής θέλω να πω και το λέγω ότι δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι πρέπει να πιεστούμε πραγματικά να εκμεταλλευτούμε και να χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο που έχουμε πλήρως στη διάθεσή μας. Έχουμε αφενός συζητήσει την έκθεση της Πεβάνς Μπερές με πρώτες αντιδράσεις. Σήμερα το προτέρημα είναι εκείνο το ότι η έκθεση είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες. Κάθε ένας, ακόμα και αν δεν κατέχει τόσο καλά τα αγγλικά, μπορεί στη γλώσσα του να διαβάσει και να εξοικειωθεί με αυτή την έκθεση. Και έτσι υπάρχει η μία ή η άλλη, ας το πω έτσι, πτυχή που μπορεί να συζητηθεί και αύριο είναι η προθεσμία που εκπνέει για την κατάθεση τροπολογιών. Και γι' αυτό θα έλεγα ότι κάθε ένας από εμά εντωμεταξύ θα, μπορεί, θα πρέπει να έχει καταλήξει στα δικά του συμπεράσματα και να έχει μπορέσει να διατυπώσει τις ε, απόψεις του για αυτή την έκθεση. Θα πρότεινα μας πολύ σύντομα να κάνεις μια εισαγωγή. Δεν χρειάζεται να είσαι εκτενέστερη, έχεις ήδη παρουσιάσει την έκθεσή σου. Κάποια λεπτά σύντομα να μας παρουσιάσεις πώς έχουν τα πράγματα. Ποιο είναι το κύριο μήνυμα της έκθεσής σου, ώστε μετά στη συνέχεια να περάσουμε στη συζήτηση. Παρακαλώ Περβάνς. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ πρόεδρε και εγώ επίσης χαίρομαι που ξαναβρίσκω εδώ τον Ότμαρ Καράσα που είναι σε καλή υγεία ε, μεταξύ μας. Η υγεία του προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις του επαγγελματικής ε, για την ε, Επιτροπή Κρίσα διότι τον χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή, όχι πως δεν μας έλειψε κατά τη διάρκεια της ενδάμεσης περίοδου. Αύριο είναι το, η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών σύμφωνα με το πνεύμα ε, νομίζω που υιοθετήθηκε. Όλες οι τροπολογίες ε, θα υιοθετηθούν από τον εισηγητή, του Σκιώδης, εισηγητές και ελπίζω να μην ξεπεράσουν ένα λογικό αριθμό. Έχετε το κείμενο σε όλες τις γλώσσες και το γαλλικό κείμενο έχει μια νέα εκδοχή διορθωμένη και καλό τους γαλλόφωνους να αναφέρονται σε αυτήν ε, το καινούριο κόμμενο που δεν μεταφράζει το fiscal με φορολογία αλλά με δημοσιονομικό. Κάτι άλλο σχετικά με τους τύπους θα ήθελα απλώ να πω ότι στην έκθεση έτσι όπως κατατέθηκε υπάρχουν ορισμένοι αριθμοί, ορισμένα στοιχεία. Για ένα λόγο που μου διαφεύγει αναφέραμε τις παραπομπές, τις αναφορές των κειμένων στα οποία παραπέμπει το κείμενο αυτό. Νομίζω ότι αυτές οι τεχνικές λεπτομέρειες θα προσθεθούν από τη γραμματεία ούτως ώστε η εργασία μας να είναι και τυπικά καλύτερη ποιότητα. Τα βασικά μηνύματα τα γνωρίζετε, είναι αυτά τα οποία συμφωνήσαμε ε, στην επανέναρξη των εργασιών μας σε αυτό το δεύτερο μέρος της θητείας μας για να επικεντρωθούμε όχι μόνο στην αναδιατύπωση αυτού του οποίου είχαμε ήδη συμφωνήσει, δεν πρόκειται να ξανανοίξουμε τα σημεία που απετέλεσαν αντικείμενο κονσένσους ε, στην ενδιάμεση έκθεση, δεν έχουμε θέμα θέματα που εξαρτώνται από νομοθετική εργασία άλλων επιτροπών δεν ε, γινόμαστε μια νέα επιτροπή Γκονζάλες αλλά ταυτόχρονα προβαλόμαστε κάπως μακρύτερα στον ορίζοντα τον κοινοβουλευτικό και με το πνεύμα αυτό μου φαίνεται ότι υπάρχουν μερικά σημαντικά σημεία σε αυτή τη νέα έκθεση. Πρώτα απ' όλα η, ο τονισμός της σημασίας να αποκατασταθεί εμπιστοσύνη και ε, το όραμα στην εγχείρημα το ευρωπαϊκό, η εμπιστοσύνη ότι μπορεί να φέρει στην συνολική συζήτηση ε, γύρω από το ευρώ σημαντικά στοιχεία και για το διεθνές νομισματικό σύστημα που παρουσιάζει σήμερα ένα διπλό μειονέκτημα που είναι ότι έρχεται σε αντίφαση δυνητική της τις ανταγωνιστικότητα ανταγωνιστικότητας των κρατών μελών και ευνοεί κερδοσκοπίες όσον αφορά τις ισοτιμίες και τις ανταλλαγές νομισμάτων, πράγμα που είναι αντίθετο προς τους στόχους μας. Άλλο σημαντικό σημείο που υπενθυμίζουμε σε αυτήν την έκθεση στην παράγραφο 31 και 32 λόγω των ανισορροπιών των εσωτερικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε πολύ επιμείνει στην πρώτη έκθεση και η συνέχεια των γεγονότων δεν ήρθε να μας διαψεύσει αλλά αντίθετα είδαμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε μία μοναδική ενιαία λύση για να αντιμετωπίσουμε όλες τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρόλο που ανήκουμε σε μια ίδια ένωση και παρόλο που ορισμένα κράτη έχουν το ίδιο νόμισμα. Δεύτερο σημείο που έχει μια διάσταση ευρωπαϊκή και στο οποίο αποδίδω πάρα πολύ μεγάλη σημασία και νομίζω ότι και οι πολιτικοί ηθήνοντες εδώ δεν έδωσαν την δέουσα σημασία. Είναι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αρκετά πλούσια ούτω ώστε μόνη τη να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους που έχει ορίσει. Και αν δεν έχουμε συνεκτικότητα, συμπληρωματικότητα και αν δεν έχουμε ένα εργαλείο σύγκρισης για να μπορέσουμε να διαρθρώσουμε ε, μια στρατηγική ευρωπαϊκή για τον προϋπολογισμό τον ευρωπαϊκό και τους εθνικούς προϋπολογισμούς αφετέρου δεν θα έχουμε καμία πιθανότητα επιτυχίας. Τηλεγραφικά κύριε Πρόεδρε, θα, για να προβληθούμε στο μέλλον αυτό που θέλαμε στο έκτο θέμα το οποίο είχαμε συγκρατήσει για τις εργασίες μας πέρα από την οικονομική διακυβέρνηση και την νομισματική για να επιμείνουμε πάνω σε πέντε σημεία τα οποία μου φαίνονται σημαντικά. Το πρώτο, ότι στις χρηματοπιστωτικές αγορές μια από τις δυσκολίες σήμερα και νομίζω ότι ο πρόεδρος και ο γενικός διευθυντής του ε, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σήμερα έχουν, ε, ομιλούν προς την ίδια κατεύθυνση. Έχουμε πολύ επικεντρώσει τις προσπάθειές μας στο θέμα της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών. Κανείς ε, δεν μιλάει για την αμφισβήτηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, αλλά η απλή παρατήρηση της σταθερότητας των χρηματοοικονομικών αγορών δεν θα μας επιτρέψει να επιλύσουμε το πρόβλημα των παγκόσμιων ανισορροπιών που οδήγησαν σε αυτή την κρίση κρίση. Η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών θα μας επιτρέψει να επανέλθουμε στην εξάντε κατάσταση του 2007, όχι να εξαλείψουμε τα αίτια της κρίσης. Θα πρέπει να σκεφτούμε, και αυτό είναι δύσκολο έργο, να σκεφτούμε μηχανισμούς που θα μας επιτρέψουν να παρακολουθούμε την βέλτιστη διοχέτευση των κεφαλαίων βάσει των μακροοικονομικών στόχων που τηρούμε που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δεύτερη σημαντική παρατήρηση είναι βεβαίως το θέμα της ικανότητας των ελεγκτών της εποπτείας να φέρουν σε πέρα στο έργο τους το είδαμε όταν επρόκειτο να οριστούν οι ελεγκτές, οι νέες αρχές, είδαμε πως υπήρχαν παρεκτροπές τις οποίες έπρεπε να ε, καταπολεμήσουμε. Τρίτο θέμα είναι ότι σε πρόπτικη, αν είμαστε συνεκτικοί με τους και συνεπίσα, με τους στόχους που ορίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός σε έναν ορίζοντα που δεν αναφέρω σήμερα θα πρέπει να αντιπροσωπεύει σημαντικότερο μέρος του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέταρτο στοιχείο, όπως είχαμε συμφωνήσει στην αρχή της δεύτερης φάσεις των εργασιών μας, να προσδιορίσουμε συγκεκριμένα σημεία για τα οποία η σημερινή συνθήκη δεν είναι υπαρκής για να μας επιτρέψει τα στάδια τα οποία χρειαζόμαστε για την ολοκλήρωση και την ενοποίηση με δυστυχώς ε, την αναγκαιότητα να ξανατονίσουμε ότι αν χρειαστεί να ξανανοίξουμε το θέμα της συνθήκης της Λισαβόνας δεν θα μπορούμε να δεχθούμε αυτό να γίνει με τους ίδιους όρους όπως έγινε σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθεροποίησης θα πρέπει να απαιτήσουμε αυτό να οδηγήσει σε μια σύμβαση όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει νέα δικαιώματα με τη συνθήκη της Λισαβόνας να συνδεθεί με τις εργασίες και τη σύνταξη αυτής της νέας συνθήκης και άλλη μια φορά εδώ αναφέρουμε μερικούς άξονες τους οποίους θα έπρεπε να ακολουθήσει αυτή η αναθεώρηση. Συμπερασματικά μπορώ να πω ότι δυστυχώς θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης που έχουν ιδιαίτερη ευθύνη επειδή είναι μέλη, επειδή μοιράζονται ένα ίδιο νόμισμα θα έπρεπε να σκεφτούν μεταξύ τους μια ενισχυμένη συνεργασία διότι είναι μια λύση την οποία δεν δέχομαι ελαφρά την καρδία. Ε, το να, αν δεν μπορούν όλοι μαζί, όλοι μαζί να κάνουμε κάτι ε, και αν αυτοί που είναι πιο προχωρημένοι είναι όμοιροι αυτών που δεν θέλουν να προχωρήσουν και που δεν μοιράζονται τις ίδιες ευθύνες εφόσον δεν έχουν την ευθύνη της επιβίωσης του ευρώ, τότε θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να σκεφτούμε όχι de facto αλλά de jure μια ενισχυμένη συνεργασία. Αυτά είναι μερικά από τα στοιχεία που σας υπενθυμίζω και που είναι η ουσία του δευτέρου σταδίου της έκθεσης που θα είναι νομίζω και το τελικό στάδιο ακόμα και λόγω της εξέλιξης της κρίσης δεν είναι βέβαιο ότι όταν θα ψηφίσουμε τον Ιούλιο για, αυτή, αυτήν την έκθεση ότι θα έχει λήξει η κρίση αλλά πάντως εμείς θα έχουμε κάνει το καθήκον μας. Ευχαριστώ πολύ, Πεβά. Θα πήγαινα πιο πέρα ακόμα, Πεβά, ότι είναι σίγουρο ότι δεν έχει περάσει ακόμα η κρίση σε σχέση με την ψήφο, ψήφιση της έκθεσής σου. Ας ελπίσουμε τα καλύτερα όμως. Φοβούμαι ότι μια ολόκληρη σειρά ετών θα μας συνοδεύει. Δεν πάω τόσο μακριά όσο ο συνάδελφός μας, ε, ο κύριος Φιλαγγελίδης, εχθές ο φιλοξενούμενος, ότι επί μια γενεά θα ε, συμβεί αυτό και θα μας συνοδεύει. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να τα ξεπεράσουμε και ο κύριος Σότμα Κάρας θα λάβει τώρα τον λόγο. Παρακαλώ. Πρόεδρε, πρώτα θέλω να ευχαριστήσω για τις, ε, τα συγχαρητήρια και τις ευχές σας. Πιστέψτε μου, Πιστέψτε με, ήταν δύσκολη η περίοδος που πέρασα. Χαίρομαι που ξαναβρίσκομαι ανάμεσά σας στο Ευρωκοινοβούλιο. Τώρα, όπου η κατάσταση είναι μια τελείως διαφορετική από ότι σε σχέση με την πρώτη έκθεση που είχε συνταχθεί τότε έχουμε καλύτερα θεμέλια πλέον στη διάθεσή μας και αυτή η βάση, αυτά τα θεμέλια που έχουμε τώρα στη διάθεσή μας δεν μας χωρίζει πια τον ένα από τον άλλο τόσο σημαντικά. Η κατεύθυνση είναι κοινή για όλους μας και πρέπει να αναμείνουμε και να δούμε τι θα γίνει με τις ε, τροπολογίες που θα κατατεθούν και με βάση αυτές τις τροπολογίες να συμπληρώσουμε την έκθεση ή να την βελτιώσουμε αν γίνεται. Είναι πραγματικά μια σαφής βάση αυτή που έχουμε και που βασίζεται στην πρώτη έκθεση, στην ενδιάμεση έκθεση και η σωστή κατεύθυνση είναι αυτή. Και μπορούν τα πράγματα να δούμε αν μπορούν να βελτιωθούν. Αυτή είναι η προσπάθειά μας, να βελτιωθούν. Δεύτερον, εμείς ως κοινοβουλευτική ομάδα θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία όπως την τελευταία φορά. Δηλαδή να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς από πλευρά της ομάδα μας που θα καταθέσουμε εξ ονόματο της ομάδας μας και αν είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει ξεχωριστά να γίνουν κάποιες ατομικές τροπολογίες αν θεωρούν τα μέλη. Αλλά όπως η συγγήτρια ήταν απόλυτα σαφής όχι μόνο σε σχέση με ατομικές τροπολογίες αλλά και σε σχέση με τις άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες θα γνωρίζουν ποια είναι η δική μας θέση ως ομάδα και ποια θέματα είναι για μας ιδιαίτερα σημαντικά. Πρόκειται για μια εμβάθυνση και συμπλήρωση λοιπόν. Το τρίτο. Το τρίτο είναι ότι θα παρακαλούσα τους άλλους σκιώδεις εισηγητές και συντάκτες τροπολογιών θα ήθελα να τους παρακαλέσω υπό το φως των τροπολογιών αυτών να βασιστούν στα θεμέλια, στη βάση της πρότασης και με βάση την εμπειρία της χθεσινής μας συζήτησης να καταλήξουμε στη σύνταξη του πίνακα ψηφοφορίας και ή δυνατών συμβιβασμών. Είναι γεγονός ότι με τις τροπολογίες που εμείς καταθέτουμε μπορούμε να πούμε εκ προημίου, θα ήθελα να πω εκ προημίου ότι πρόκειται για τροπολογίες λοιπόν που αποσαφηνίζουν ότι δεν πρόκειται για νομοθετικής, ε, νομοθετικού χαρακτήρα έκθεση. Αν ήταν νομοθετικού χαρακτήρα έκθεση, πολλές από αυτές τις τροπολογίες δεν θα μπορούσαμε να τις καταθέσουμε. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να είναι αυτή μια έκθεση η οποία πρέπει να είναι μια έκθεση που θα αποσαφηνίζει, θα διευκρινίζει ότι εμείς με αυτή την έκθεση δεν κάνουμε μια καθημερινή πολιτική από μέρα σε μέρα καθημερινά και οικία, αλλά θαραλέα κάνουμε το βήμα προς το μέλλον με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, μακροπρόθεσμη προοπτική προς την κατεύθυνση στην οποία θέλουμε να κινηθούμε. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι και σε εμά αλλά και στις άλλες ομάδες. Πολλοί συνάδελφοι που σε κάποιες διατυπώσεις ε, τροπολογιών ή τοποθετήσεων θα πούν «Μα πώς θα τα εξηγήσω αυτά στους ψηφοφόρους μου» Λέω όμως ότι η αλήθεια είναι κάτι αδιαμφισβήτητο, κάτι ανίκητο. Και αν δεν ξεκινήσουμε εμείς τότε τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση και για τις μακρόχρονες προοπτικές αν δεν τα εξηγήσουμε όλα αυτά και δεν προχωρήσουμε τότε στους πολίτες μας δεν θα μπορέσουμε τους πολίτες να τους κερδίσουμε για βράχη πρόθεσμα μέτρα προσωρινού χαρακτήρα. Γι' αυτό παρακαλώ όλους όχι μόνο την καθημερινή δουλειά από πλευράς πολιτικού, πολιτικής να εξετάσουν και τα σήμερα ήδη κατανοητά, να μην αντιμετωπίσουν αυτή την κατεύθυνση, αλλά το αναγκαίο για την Ευρώπη στο μέλλον. Και αυτό που είναι αναγκαίο για την Ευρώπη για το μέλλον είναι για τους πολίτες μας το πιο χρήσιμο και για τα κράτη-μέλη το πιο χρήσιμο. Είδαμε ρητά και κατηγορηματικά ότι μια νομισματική ένωση αυτών των διαστάσεων με αυτές τις εξελίξεις με ένα προϋπολογισμό 1% δεν μπορεί να είναι αξιόπιστη μια τέτοια ένωση με τέτοια μέσα οικονομικά. Δεν θέλαμε όμως να ασκήσουμε μόνο επικρίσεις, εντάξει. Πρέπει μακροπρόθεσμα να πούμε ποιοι είναι οι στόχοι μας, μακροπρόθεσμα στην πολιτική μας. Δεύτερο, είναι φυσικά σαφές ότι όλα αυτά με τις συνεισφορές των κρατών μελών αποκλειστικά δεν μπορούν να καλυφθούν χρηματοοικονομικά. Και γι' αυτό η συζήτηση για τους ίδιους πόρους πρέπει να ξεκινήσει και να προαχθεί. Και εδώ ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε κοινέ διατυπώσεις μέσω της έκθεσής μας. Και έτσι και εδώ θα πρέπει οι σκιώδεις εισηγητές και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, οι Ευρωβουλευτές, να δημιουργήσουν διασταυρούμενες τοποθετήσεις αν δεν θέλουμε να διακυβευτεί η αξιοπιστία της κοινοβουλευτικής μας θέσης και τοποθέτησης. Και εδώ λοιπόν έχουμε ένα έργο συντονισμού στο οποίο πρέπει να προβούμε και να διασφαλίσουμε. Είδαμε ότι δεν έχουμε επαρκείς ευρωπαϊκές αρμοδιότητες ώστε πολιτικά να είμαστε αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση της κρίσης και μάλλον διακυβερνητικά επίπεδα και εθνικά επίπεδα δραστηριοποιούνται για να δοθούν οι απαντήσεις που χρειάζονται σήμερα. Όμως από την άλλη πλευρά είδαμε ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε κρίσεις και παρόλα αυτά αυξάνονται τα κρατικά χρέη. Γι' αυτό η μείωση των ελλημάτων. Για μας είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο και σπουδαίο. Και χωρίς μεταρρυθμίσεις, χωρίς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, χωρίς ανταγωνιστικότητα, χωρίς ανάπτυξη και απασχόληση, χωρίς την ενίσχυση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς, χωρίς την υλοποίηση μιας ταμιακής εξυγίανσης ώστε να δούμε τι είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε και πόσα χρήματα χρειαζόμαστε για να τα πετύχουμε όλα αυτά και με ποια μέτρα θα μπορέσουν όλα αυτά να γίνουν σε αυτή την πλευρά μπορεί η έκθεση ακόμα να ενισχυθεί, να ενδυναμωθεί και να τονωθεί. Έχουμε προβλήματα φυσικά με τον εναρμονισμό των φορολογιών, των ε, φόρων. Το θέμα του εναρμονισμού ή το θέμα το φορολογικό δημιουργεί τελείως διαφορετική προοπτική για την αναγκαία αυτή εξέλιξη της Ευρώπης και την εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη στη δημοσιονομική πολιτική, στην οικονομική πολιτική, στην ε, φορολογική πολιτική, στην κοινωνική πολιτική, στην πολιτική για την παιδεία, εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά χρειαζόμαστε επίσης και τον ανταγωνισμό μεταξύ των βέλτιστων. Δηλαδή, ο εναρμονισμός ε, πρέπει να δούμε αν συνοδεύεται από την προώθηση και του ε, ανταγωνισμού και να μην ε, παρακολεί μια κατεύθυνση η οποία θέλουμε να ακολουθηθεί. Και γι' αυτό ο ε, εναρμονισμός απόλυτος ο εναρμονισμός δεν σημαίνει κατάργηση της Ευρώπης ε, ο ανταγωνισμός δεν σημαίνει εξίσου αρνητικές εκτόσεις για την Ευρώπη και γι' αυτό θα πρέπει να καταλήξουμε σε αυτή, καταλήξαμε σε αυτή την ευρεία συνένεση ως ομάδα έχουμε το στόχο να εκφράσουμε τις δικές μας θέσεις ε, για το μέλλον φιλόδοξα και να μην αναζητήσουμε τον ελάχιστο κοινό παρονόμαστη και χαίρομαι και προσβλέπω στη συζήτηση που θα διεξαχθεί για να συμπληρωθεί και να τονωθεί η έκθεση, να ενδυναμωθεί ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ για το έργο που επιτελέσατε. Βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερη θέση σήμερα από ό,τι στο παρελθόν και γι' αυτό δεν χρειάζεται μόνο να συντονιστούμε, αλλά μπορούμε από κοινού να κάνουμε αυτά επόμενα βήματα προς τα εμπρός, προς το μέλλον και έτσι να δείξουμε ότι το έργο μας το παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά, με ιδιαίτερη σοβαρότητα δρούμε και το πρόγραμμα εργασίας για όλους, για το μέλλον, με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζεται. Σας ευχαριστώ. Äh, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα μεθοδολογίας, Επιβεβαιώνω και εγώ ότι η ομάδα των Σοσιαλιστών και των Δημοκρατών, και Δημοκρατών θα παρουσιάσει, θα υποβάλει τροπολογίες που θεωράει ότι είναι χρήσιμα να ενταχθούν για να ενισχυθεί η έκθεση της Περόνς Μπερές. Έχοντας ε, προηγουμένως βέβαια ε, κάνει εντελεχή συζήτηση στους κόλπους της και έχοντας για πρώτη σύνθεση των θέσεων αυτών, Ακριβώ για να ενισχυθούν τα επιχειρήματα και να ενισχυθεί η εργασία, όπως είπαμε, που είχαμε δεσμευτεί να επιτελέσουμε στην τελευταία συζήτηση της Επιτροπής μας. Σε ό,τι αφορά την ουσία, νομίζω ότι η έκθεση της Περόνς έχει πάρα πολλές θετικές πτυχές και εξαιρετικά σημαντικές. Θα ήθελα εντάχει να υπογραμμίσω δύο στοιχεία. Το ένα είναι η ικανότητα που όλοι μαζί, αν θα το ρημάσουμε κατά τη διάρκεια της μακραυτής περίοδου, να εντοπίσουμε συγκεκριμένους στόχους ανάληψης πρωτοβουλειών. Για παράδειγμα, επιβεβαίωση ανάμεσα στις προτεραιότητες της έκθεσης αυτής ...την ε, πρωτοβουλία ενεργητικών ε, πολιτικών και σε θέματα επίσης ε, ένταξης και μετανάστευσης. Πρέπει δηλαδή να αντιμετωπίσουμε και κάποια κατεπήγοντα ζητήματα με πρόθεση να δούμε πιο μακριά, όπως μόλις ζήτησε και ο συνάδελφος Κάρας. Είναι προφανές ότι τα δραματικά γεγονότα της Ιαπωνίας αφενός και η κρίση της ε, Νοτιού Μεσογείου από την άλλη μας ε, παραπέμπει σε διαφορετική ε, αντιμετώπιση του ενεργητικού, του θέματος ενέργειας και της εξέλιξης τεχνολογιών. Είπαμε ότι με πολύ ε, μεγάλη, αν θέλετε, καθυστέρηση, ότι πέρα από τα κατεπήγοντα, τα οποία έχουν, κατεπήγοντα ζητήματα που έχουν εμφανιστεί, συνιστά μία από τι ε, θεμελιώδεις και πρώτες, ε, αν θέλετε, πιο βασικές, βασικά προαπαιτούμενα για την ε, πολιτική, την ευρωπαϊκή πολιτική τη επόμενη δεκαετία. Το ίδιο ισχύει και με τα θέματα τη μετανάστευση. Αντιμετωπίζουμε εκατοντάδες χιλιάδες άτομα που φεύγουν από τη χώρα του που έρχονται προς την Ευρώπη. Άρα πρέπει με μεγάλη αποτελεσματικότητα και πολύ καλή στόχευση να αντιμετωπιστούν τα κατεπήγοντα αυτά. Αλλά η Περβάνς επαναλαμβάνει στο θέμα της μετανάστευσης και την απέτηση του να υπάρχουν κοινέ πολιτικές για την Ευρώπη σε ό,τι αφορά την μετανάστευση. Γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη υποφέρει από πολύ μεγάλη δημογραφική ανισορροπία και για να επιτευχθούν οι στόχοι τους οποίους έχουν θέσει εδώ, θα είναι απαραίτητο να έχουμε ανάμεσά μας πάρα πολλού που θα έχουν γεννηθεί σε άλλη πλευρά του κόσμου και που θα αποφασίσουν να έρθουν να, δουλέψουν, να ζήσουν και να δουλέψουν σε εμά. Οι πολιτικέ μετανάστευση λοιπόν δεν θα πρέπει ποτέ να γίνονται αντιληπτέ σαν πολιτικέ του κατεπήγοντο, αλλά θα πρέπει να είναι ένα απόσπαστο κομμάτι των ε, στρατηγικών επιλογών που κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν μπορώ παρά να συγχαρώ και, γιατί, και να συμφωνήσω με την δεύτερη παρατήρηση που γίνεται. Πιστεύω ότι πολύ, πολύ σωστά περιγράφηκε στην έκθεση της Περβάνς και συμφωνώ και τονίζω ότι οι τροπολογίες του κατεθούν δεν θα αλλάξουν το όλο σκεπτικό της ηγήτριας. Εάν δεν τους, ε, εάν τις αποδεχθεί θα τις αποσύρουμε. Αυτό θέλω να πω λοιπόν ότι είναι κινούμενοι με την απέτηση να υπάρχουν επαρκείς λύσεις που προκύπτουν από την ε, χρηστή διακυβέρνηση, από την governance στην ευρύτερη, αλλά προκειμένου να υπάρξει και ένα θαραλέο βήμα προς την πολιτική ένταξη, τόσο οικονομικής όσο και θεσμικής, Εάν δεν υπάρξει κάτι τέτοιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση διακινδυνεύει να αντιμετωπίσει πάρα πολύ μεγάλε δυσκολίε στο μέλλον. Πέραν και εκτό τη όλη κρίση. Δηλαδή, το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση έγκυται στην ικανότητά τη να ενισχύσει όλου του μηχανισμού ε, ολοκλήρωση. Ξεκινώντας βεβαίως ε, άμεσα σε αυτού που αφορούν την άμεση οικονομική νομισματική πολιτική μπορούσαμε να είχαμε ολοκληρώσει την εργασία σε αυτήν την επιτροπή με πάρα πολλού τρόπου, δίνοντα απλώ παρατηρήσει μα, υποβάλλοντα κάποιε προτάσει, υπογραμμίζοντα ε, τα σημεία τη ανάλυση πάνω στο γιατί μα έφτασε και μα έπληξε η κρίση. Ποιε ήταν τα και ποιε ήταν οι κύριε επιπτώσει, ανεταιρικέ επιπτώσει κοινωνικού χαρακτήρα και να σταματήσουμε εκεί. Ανταυτού κάνουμε μια επιλογή που είναι απόλυτα συνειδητή, αλλά κατ' εμέ είναι και μοναδική πολιτικά σωστή λύση Δηλαδή να υποδείξουμε ποιο μπορεί να είναι το μέλλον της Ευρώπης, μιας μεγαλύτερης ολοκλήρωσης, δηλαδή καινοποίησης. Βέβαια, ε, σε αυτή την επιτροπή, δεν επαφή σε αυτή την επιτροπή να υλοποιήσει και να κάνει αυτή την αλλαγή. Δεν πρόκειται για νομοθετικό κείμενο, αλλά ε, προγραμματικών δηλώσεων. Όμως, τα συμπεράσματα μιας επιτροπής, σαν τη δική μας, καλά στοχευμένη σύγχυση πάνω στην οικονομική νομισματική και κοινωνική κρίση, το, τον κατακλείδη συμπέρασμα, όπως είπα, είναι πολιτικό. Και πιστεύω άμεσα όχι μόνο σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας και εργασίας, αλλά και στο τι θα προκύψει σε σχέση με τις συζητήσει που έλαβαν χώρα εδώ και δύο χρόνια. Το μέλλον τη Ευρώπη περνά από την απόφαση των κρατών μελών να δώσουν στην ίδια την Ευρώπη μεγαλύτερη συνοχή και δει μια δομή που θα ενδυναμώνει την θεσμική της ε, δομή, ξεκινώντας ακριβώς και με βάση αυτή την πολιτική βούληση, όπου τα διάφορα πολιτικά κόμματα στις διάφορες χώρες και οι κυβερνήσεις που ανάλογα εκπροσωπούν τα πολιτικά αυτά κόμματα, ανάλογα με το πνεύμα κάθε φορά που διέπει την συμπολίτευση, θα τα υλοποιήσουν. Από εκεί θα περάσει η Ευρώπη και αυτός είναι ο στόχος μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ήδη συνεχάριν την κυρία Μπερέσα για την εργασία της. Μπορώ να το κάνω και πάλι και να το επαναλάβω και πάλι. Αλλά νομίζω ότι εφόσον μιλούμε για κρίση θα έπρεπε καμιά φορά να αναφέρουμε ότι η Ευρώπη βρίσκεται ακόμα εκεί, η Αμερική βρίσκεται ακόμα εκεί. Όταν είχαμε κρίση στη δεκαετία του 20 του 30 ξέραμε τι συνέβαινε, ξέραμε ακριβώς περί σε πρόκειται. Τώρα όχι. Αν θέλουμε ε, οι ε, πολίτες να πιστεύουν στην Ευρώπη θα έπρεπε να πούμε και κάτι το θετικό, όχι να προσπαθούμε πάντοτε να εξηγήσουμε γιατί το ποτήρι είναι μισό άδειο. Θα πρέπει καμιά φορά να τους λέμε ότι είναι και μισό γεμάτο το ποτήρι. Ε, πολύ συχνά εκπλήσουμε με αυτά που κάνουμε και με αυτά που επιτυγχάνουμε. Ναι, ναι, όντως. Και πιστεύω ότι ε, καμιά φορά είμαστε πάρα πολύ υπερβολικά αρνητικοί. Αν είμαστε εμεί λοιπόν τόσο αρνητικοί, πώς να είναι θετικοί οι πολίτες. Στην πρώτη έκθεση ε, στο συμπέρασμα ήταν περισσότερη Ευρώπη. Συμφωνώ, είμαι πολύ ευρωπαϊστής και καμιά φορά όταν προσπαθώ να συνηγορήσω υπέρ της Ευρώπης στην χώρα μου, ορισμένοι λένε ότι είμαι ουτοπιστής, ότι είμαι τρελός. Ε, πρέπει να δίνουμε τις σωστές απαντήσεις δεν μπορούμε όμως σε κάθε ερώτηση να απαντάμε ε, με, θα λυθεί το θέμα με περισσότερη Ευρώπη. Δεν μπορούμε πάντοτε να ζητούμε περισσότερη Ευρώπη. Στην πόλη μου οι πολίτες ε, θέλουν πιο ισχυρούς πολιτικούς, εθνικούς ε, και τοπικές αρχές στην εθνική αρένα. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πιο προσεκτικοί. Κυρία μου, έχουμε περίπου 50-60 τροπολογίες μέχρι τώρα. Θα έπρεπε να μιλήσετε με τον πρόεδρο γι' αυτό. Προσπαθούμε, αλλά μερικές τροπολογίες ε, είναι δευτερεύουσες αλλαγές. Να εξηγήσω. Μερικές ε, τροπολογίες αντικαθιστούν μία λέξη με μία άλλη. Αυτό προσπάθησα να πω. Είναι ασήμαντες αλλαγές. <coughs> Και θα υπάρξουν και ατομικές τροπολογίες. Θα ήθελα όμως σύντομα να πω που έχουμε μερικές ανησυχίες. Θα θέλαμε να μιλάμε για στενότερη ε, συνεργασία για την φορολογία. Μπορούμε ε, να εγκρίνουμε το ευρύτερο όρομα, αλλά όχι σήμερα όταν αν θέλουμε να έχουμε ένα ταμείο, ένα ευρωπαϊκό οικονομικό, μια οικονομική οντότητα, ίσως είναι υπερβολικό. Ένα μέρος της ομάδας μας σκέφτεται ότι τα ευρωομόλογα δεν θα σώσουν το, την Ευρώπη, δεν θα λύσουν το πρόβλημα της Ευρώπης, αλλά έχουμε στην ομάδα μας μερικές διαφορετικές απόψεις και ίσως να δούμε ε, μερικά αποτελέσματα. Θέλουμε ένα μηχανισμό για το ξεκαθάρισμα, για να καθαρίσουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Δεν νομίζω ότι αναφορά στην Deutsche Börse και στο Αμερικανικό χρηματιστήριο χρειάζονται εδώ ε, κυρίως όταν ε, το Nasdaq, MEX ε, θέλουν επίσης να θεωρηθούν χρηματιστήρια παρόλο που απορρίφθηκαν αλλά μπορεί να έχουν καλύτερο επίπεδο αύριο κυρία μου. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες μελέτες σχετικά με την παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση. Κατανοώ τις προτάσεις σας αλλά πρέπει να ξέρουμε περισσότερα και όπως είπαμε προηγουμένως το G20 είναι και, και θα μπορούσε να είναι ένα βασικό ε, σώμα που λαμβάνει αποφάσεις. Νομίζω ότι οι στόχοι της ε, χιλιετίας πρέπει ε, να υλοποιηθούν και είναι μόνο τέσσερις χώρες που τηρούν αυτά τα κριτήρια της χιλιετίας και τους στόχους της χιλιετίας. Δεν ξέρω ότι θα έχετε κάτι να πείτε επιστρέφοντας στις πρωτεύουσές σας και στα εθνικά σας κοινοβούλια. Θα πρέπει να αρχίσουν ε, τηρώντας τις δικές τους υποχρεώσεις ε, και δεσμεύσεις και να μην ε, στρέφονται στην Ευρώπη. Όπως είπαμε επίσης, πιστεύουμε ότι η Μαριομόντι είναι πάρα πολύ καλός και ο πρόεδρος είπε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο Μάριο Μόντι. Ε, προσπαθήσαμε να το εξηγήσουμε αυτό σε μερικές τροπολογίες. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ ε, νομίζω ότι θα αποκλίνουμε από τις προτάσεις σας. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιλύσουμε πρώτα τα προβλήματά μας προτού να πούμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα. Νομίζω ότι είναι κατάλληλο, ότι κατάλληλο είναι πολύ πιο καλή λέξη, καλή διατύπωση και υπάρχουν μερικά κονδύλια που κακοχρησιμοποιούνται ήδη στον προϋπολογισμό. Όπως είπα προηγουμένως, νομίζω ότι το τελευταίο θέμα ασχοληθήκαμε με, με το, την τελευταία περίοδο ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό στο Κοινοβούλιο και ε, φερθήκαμε κακώς, γιατί νομίζω ότι το προϋπολογισμός ο κοινότικό θα έπρεπε να έχει μέτρα λιτότητας και την περασμένη εβδομάδα πήραμε μερικές αποφάσεις που δεν ήταν ε, φρόνιμες σχετικά με τον προϋπολογισμό, σχετικά με την κυβερνητική δραστηριότητα και την Επιτροπή. Συμφωνούμε πλήρως μαζί σας, κυρία μου, και ενισχύσαμε μάλλον μερικές από τις προτάσεις σας πολιτική μεταναστευτική που αναφέρθηκε εδώ. Συμφωνώ πλήρως και νομίζω ότι πρέπει εδώ να είμαστε ε, πιο δυνατοί, πιο ε, αυστηροί. Ε, υπάρχουν λίγες χώρες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσει Λαμπεντούζα και αυτό είναι ντροπή. Όνειδος. Τώρα έχουμε μια δημοκρατική επανάσταση στην Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή και το γιορτάζουμε αυτό, το επικροτούμε, αλλά δεν θέλουμε να έρθουν εδώ οι πολίτες των χωρών αυτών. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό και δεν είμαστε πρόθυμοι να αλλάξουμε την εμπορική μας πολιτική. Αν θέλουμε να είμαστε ένα σοβαρό εταίρος ε, στην γειτονιά μας θα πρέπει να αλλάξουμε γρήγορα και σημαντικά. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της ομάδας ALDE. Ευχαριστώ. The Ευχαριστώ κυρία, κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα λίγο, αλλά μόλις ήρθα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η ομάδα μας ε, είχε κάποιες δυσκολίες με την έκθεση αυτή υπό την έννοια ότι κάποιες από τις προτάσεις ε, ίσως δεν είναι, αν θέλετε, αναπάντεχες. Συχνά έχουμε δυσκολίες με θέματα που προτάσει η κυρία Μπέρες, όπως θέματα εναρμόνισης φορολογίας και θέματα που αφορούν τον κοινοτικό προϋπολογισμό, κατά πόσο είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος. Φοβάμαι ότι η ομάδα μας πιστεύει γενικά ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι όσο δυνατόν μικρότερος και που δεν είναι να μην αυξηθεί. Και σε ό,τι αφορά τα θέματα εναρμόνισης φορολογίας, προφανώς πιστεύουμε σε μεγαλύτερο συντονισμό των φορολογιών, που είναι τελείω διαφορετική ορολογία από αυτή που χρησιμοποιείται στην έκθεση αυτή και στην οποία δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη διαφοροποίηση μεταξύ των παικτών εντό και εκτό Ευρωζώνη σε κάποια σημεία τη έκθεση και το επισημαίνουμε αυτό τροπολογίε τροπολογίες οποίες καταθέτουμε. Και σε σχέση με τα ευρωομόλογα θα προτιμούσαμε να είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκείνη που θα αναλάβει κάποια διερεύνηση των επιπτώσεων που θα μπορούσε να έχει η έκδοση ευρωμολόγων. Έχω πολύ μεγάλες ανησυχίε σε σχέση με τις χώρες με πιστοληπτική ικανότητα τριπλού α που θα επιδοτεί μέσω ευρωμολόγων άλλες χώρες με πολύ χαμηλότερη πιστοληπτική ικανότητα και πρέπει να το θεωρούμε το ιερό δισκοπότηρο αυτό. Κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας είναι να ζητούμε να συμβούν ε, κάποια πράγματα σε σχέση με, τα, με, με θέματα αν θέλετε, του εξωτερικού εμπορίου των νομισματικά συστήματα. Εκεί που δεν έχουμε έλεγχο, όπω το πόσον η Κίνα θα αποδεχθεί να κρατήσει αυτό το νόμισμα με κάποιο άλλο ή κατά πόσον οι ΗΠΑ θα παραμείνουν στο νόμισμά του να είναι το παγκόσμιο. Άρα θα συμφωνούσαμε να παραμείνουμε σε θέματα αμυγό Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι υπό τον έλεγχό μα. Και κινούμαστε τώρα σε κάποια πιο θετικά σημεία. Πιστεύουμε ότι η στρατηγική Ευρώπης 2020 είναι ε, ένας πύχης στον οποίο μπορούμε να κατατείνουμε και υποστηρίζουμε κάποιε από τι προτάσει που περιλαμβάνονται εδώ. Συνολικά θεωρούμε ότι είναι πολύ θετικό ο τόνο όλη τη έκθεση και υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία ίσονο σημασία που θα μπορούσα να διαφωνούμε, αν θέλετε. Σε ό,τι αφορά την ε, υποδομή και την, ε, αν θέλετε, παγίωση, δεν πρέπει να αναφέρουμε συγκεκριμένε εταιρείε με δεδομένα τη ρευστότητα τη αγορά, αλλά ίσω να, να επεκτείνουμε το θέμα στην, ε, αν θέλετε, ενδεχομένω συγχώνευση ή ενοποίηση ευρύτερων φορέων μεγάλων ε, εταιριών. Πάντως ευχαριστώ να υποστηρίξουμε την έκθεση. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι καινούριο αυτό στην κυρία Πέρες σε σχέση με θέματα στα οποία γενικά συμφωνούμε, άσχετα να έχουμε κάποιε διαφορετικέ διαφωνίε. Κύριο κύριος παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καθώ τελειώνουμε πια, αναρωτιέμαι για άλλη μια φορά τι θέλουμε να κάνουμε. Πώ θέλουμε να καταγραφεί στην ιστορία η έκθεση τη Επιτροπής κρίση, με βασική συγγήτρια την κυρία Μπερέζ, με πρόεδρο τον κύριο Κλίνς και παρόντες εδώ και συμμετέχοντε εμά του υπολείπου. Και το λέω αυτό κύριε Πρόεδρε γιατί συμφωνώ με το σχόλιο που κάνατε από τη χθεσινή ακρόαση, από την παρουσίαση εν πάση περιπτώσει της έκθεσης Αγγελίδη που εκτός των άλλων από τα ερωτήματα που του θέσαμε και που μας έδωσε ειλικρινείς απαντήσεις διέκρινα ότι μεταξύ του να φτιάξει ο κύριος Αγγελίδης και η Επιτροπή μια έκθεση που να συμφωνήσουν όλοι, διάλεξε το δρόμο να γράψει μια έκθεση που να τα λέει τα πράγματα όπως είναι. Και όπως θυμόσαστε όσοι τα χτες, υπήρξαν πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Αναρωτιέμαι λοιπόν, θα πριτανεύσει και στην τελική εκδοχή της έκθεσης η λογική που πριτάνευσε και σφράγισε την ενδιάμεση έκθεση, δηλαδή όσο μπορούμε να συμφωνήσουμε και αυτό είναι το μείζον και όχι κατά την άποψή μου όπως την έχω εκφράσει αρκετές φορές να πούμε πράγματα που να έχουν ε, και να στηρίζονται στην πραγματικότητα. Εν πάση περιπτώσει ε, ε, την αρχική μας γνώμη κυρίως όσο αφορά το σκέλος των διαπιστώσεων για την έκθεση της κυρίας Μπερέζη, την είχα πει στην προηγούμενη πρώτη συζήτηση που κάναμε θα καταθέσουμε κι εμείς τροπολογίες δυστυχώς θα θέλαμε να ήταν λιγότερες στον αριθμό που είπε και ο, κύριος, ο φίλος ο κύριος Σμιθ περίπου 50 τροπολογίες θα κοιτάξουμε να τις κάνουμε και λιγότερες για να μην ταλαιπωρούμε την εισηγήτρια και όλους εμάς αλλά θεωρούμε, ε, θεωρούμε επιβεβλημένο να τις καταθέσουμε αυτές τις τροπολογίες γνωρίζοντας ότι ενδεχομένω σήμερα δεν βρίσκουν μια ευρύτερη υποστήριξη αλλά ε, θεωρούμε ότι πρέπει να εξαντλήσουμε τη συμβολή μας σε αυτόν τον προβληματισμό και επιτρέψτε μου να πω ας μείνουν ως ένα καμπανάκι για κάποια πράγματα που δεν θα ήθελα να συμβούν διότι εγώ πιστεύω κύριε Πρόεδρε δεν είμαι τόσο αισιόδοξο όσο εσείς πάλι θα επικαλεστώ τον συμπατριώτη μου τον κύριο Αγγελίδη νομίζω ότι η κρίση δεν έχει ξεπεράσει και θα σας έλεγα αγαπητοί συνάδελφοι ε, εξαρτάται τώρα τι λέμε κρίση διότι αν κοιτάξει κανείς ας πούμε το ρυθμό ανάπτυξης της Γερμανίας δεν βλέπει κρίση. Αν κοιτάξει όμως ότι εδώ μετά την Ελλάδα είχαμε την Ιρλανδία, έχουμε την Πορτογαλία και ενδεχομένως και άλλες χώρες λόγω δημοσίου ελλείμματος και χρέους δεν μπορούν να το ελέγξουν μπαίνουν στο μηχανισμό και αυτή η διαδικασία και η ηφαισιακή διαδικασία απειλεί και άλλες χώρες τότε πρέπει να μιλάμε για κρίση. Κρίση, κρίση είναι μόνο κρίση του Νότου. Δεν θέλω να σας κουράσω, την τελευταία παρατήρηση την είπα απλώς για να σας πω κάποιες νήξεις ε, στις τροπολογίες που θα καταθέσουμε στο σκέλος τι θα θέλαμε να είχε. Ή αν συμφωνήσουμε και περάσουν τόσο το καλύτερο στο σκέλος ε, των διατυπώσεων, ε, ε, των αρχικών διαπιστώσεων είχα πει τη γνώμη μου. Εδώ έχει σωστές διατυπώσεις η έκθεση και διαπιστώσεις. Στις προτάσεις διακρίνω σε ορισμένες περιπτώσεις μια σαφή διατύπωση σαν να φοβάται η συγγήτρια, επιτρέψτε μου την έκφραση, γιατί δεν ξέρει και τις αντιδράσεις όλων ημών. Και τέλος υπάρχει και άλλη κατηγορία προτάσεων που είναι θετικές αυτές καθεαυτές, αλλά η εισήγηση σέβεται δυστυχώς για μένα τα περιοριστικά πλαίσια που τις αποδυναμώνουν. Ε, δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Δύο-τρεις νήξεις θα κάνω για να πάρετε μια γεύση των τροπολογιών. Την πρώτη ήδη την υπενήχθηκα από τις προηγούμενες παρατηρήσεις. Θα θέλαμε η έκθεση να λέει ότι η κρίση χρέου συνιστά, που σήμερα αντιμετωπίζουν ορισμένε χώρε έντονα, συνιστά ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Και επομένως η αντιμετώπιση του απαιτεί μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει κοινοτικοποίηση του μέρους του χρέους για να εξασφαλιστεί μια δίκαιη λύση. Δεύτερο, θα θέλαμε η έκθεση να αναγνωρίζει ότι λόγω της ύφεσης της υψηλής ανεργίας και της πτώσης των εισοδημάτων, ένα μέρος του ιδιωτικού χρέους έχει μετατραπεί σε δημόσιο. Έτσι το τελευταίο αυξάνει λόγω και της ανάγκης στήριξης και εξυγείας των τραπεζών, είπαμε αρκετά και για τις Αμερικάνικες τράπεζες χθε, και επομένως ως τέτοιο πρέπει, και ως τέτοιο πρέπει να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το τριπλό πρόβλημα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν θέλω να σας κουράσω εδώ. Θα θέλαμε τρίτον να ε, αναγνωρίζετε ρητά ότι η πλήρης απασχόληση είναι πρωταρχικό στόχος στην οικονομική, πρωταρχικός στόχος της οικονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχετικές ευαισθησίες έχω ακούσει από την εισηγήτρια. Θα θέλαμε η δημοσιονομική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδιώκει και σταθεροποιητικό αλλά και αναπτυξιακό ρόλο ε, δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, απλώς μια τελευταία ανοίξη επειδή άκουσα κάτι στην παρουσίαση. Θα πρέπει να αναγνωρίζετε ότι η ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, μπορεί να έχει αποσταθεροποιητικές συνέπειες και επομένως πρέπει να υπάρξει μια, ένα πανευρωπαϊκό σύστημα εγγύηση καταθέτεων καταπολέμησης διασυνοριακής φοροδιαφυγή. Κάτι λέει η έκθεση, θα το δώσουμε ίσως με σαφή τρόπο. Αυτές είναι οι βασικές μας παρατηρήσεις ε, ορισμένες από τις βασικές μας παρατηρήσεις και βασικές μας σκέψεις. Θα τις δώσουμε πιο αναλυτικά με τροπολογίες. Μια τελευταία παρατήρηση. Η έκθεση κάποια στιγμή πρέπει ή θα θέλαμε να διαβαστεί από τους Ευρωπαίους πολίτες. Όμως ταυτόχρονα αναδεικνύει βέβαια διακηρυχτικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται πάνω στις δημοκρατικές αρχές. Και αυτές, τις αρχές της νομιμοποίησης, αυτές το τελευταίο διάστημα περιορίζονται. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το σύμφωνο για το ευρώ πλάς, αλλά εν περιπτώσει η ιδέα, εγώ το επαναλαμβάνω, ενός πανευρωπαϊκού ή εθνικών δημοψηφισμάτων επικύρωσης του συμφώνου για το ευρώ ή της τροποποίησης της συνθήκης στο άρθρο 136 από ό,τι ξέρω ή εν πάση περιπτώσει ας βρεθεί ένας τρόπος να μιλήσουν οι πολίτες σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Κάτι θα μπορούσε να πει ως προς αυτό και η έκθεσή μας. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Äh, Ευχαριστώ Νίκο. Ο, τώρα ο Φρανκ Έγκερ, παρακαλώ. Και μετά ο κύριος Σάντσες Περσέδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα, ε, θα πω δύο λόγια στα αγγλικά, διότι κυρίως είναι μια αντίδραση αυτή σε αυτά τα οποία προανέφερε ο Όλε Σμιτ και για τον τρόπο με τον οποίο τα είπε ένα από τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε είναι μπορεί η απάντηση για όλα να είναι περισσότερη Ευρώπη. Δεν πιστεύω ότι ισχυρίζεται κανείς κάτι τέτοιο. Αν θέλουμε να καθαρίζεται ο δρόμος μας δεν μπορούμε να λέμε περισσότερη Ευρώπη για να καθαριστεί. Είναι όμως σαφές ότι σε αυτή τη χώρα δεν είναι πολλές δρόμοι καθαροί γιατί δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι αρμόδιοι για τον καθαρισμό. Και έτσι λοιπόν το περισσότερο, ε, περισσότερη Ευρώπη δεν είναι μια δήλωση, ένα αίτημα, μια απέτηση που αντικαθιστά την πιο αποτελεσματική εθνική το, περιφερειακή ηγεσία, αλλά είναι η μόνη απάντηση στα ερωτήματα που αντιμετωπίζει η δική μα Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Εμεί δεν αντιμετωπίζουμε το θέμα του καθαρισμού των δρόμων. Δεν αντιμετωπίζουμε το θέμα του ποιο θα αντικαταστήσει τι λάμπε ε, στα φανάρια που φωτίζουν τον δρόμο. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τον καθαρισμό δασών. Πρέπει όμω να καθαρίσει η ατμόσφαιρα από αυτά τα οποία την έχουν επιβερύνει τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Και αυτό κανένα κράτο μέλο δεν μπορεί να το πετύχει μόνο του <clears throat> και πάρα πολλά άλλα κράτη παγκόσμια υπάρχουν που εξακολουθούν και λειτουργούν σε ε, εθνική, με εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα και το ζουν καθημερινά εις βάρος τους ότι δεν τα καταφέρνουν. Διερωτώμε λοιπόν πώς δεδομένων όρων αυτών των αιτίων και των καταστάσεων και για το ότι έχει αποδειχθεί χωρίς να μπορεί να υποκατασταθεί πλέον ότι το μόνο πρότυπο ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που γνωρίζουμε πρέπει να ολοκληρωθεί για να καταλήξουμε στην επίλυση των προβλημάτων μας. Ή θα σταυρώσουμε τα χέρια μας και θα δούμε το τι θα γίνει αφήνοντας τα πράγματα να διολυστήσουν. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι 10 χρόνια από σήμερα, διότι χρειάστηκαν 10 χρόνια να φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση. Δεν είμαι βέβαιος όμως ότι μετά από 10 χρόνια δεν θα καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου η κανονική οδός επικοινωνίας για τους Ευρωπαίους θα έχει ξαναγίνει πιο αποτελεσματική από ό,τι ε, είναι σήμερα. Και τώρα οι ψηφοφόροι, η κοινή γνώμη έχει κάποια αντίρρηση για περισσότερη Ευρώπη. Δεν έχω ακούσει επιχειρήματα υπέρ αυτής της θέσης, ούτε έχουμε κάποια τεκμήρια και αποδείξεις υπέρ. Και γιατί συνεχίζουμε να ζητάμε συγγνώμη για το ότι υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι υπάρχουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές. Το γεγονός είναι ότι οι ψηφοφόροι και οι κοινοί γνώμοι, οι πολίτες μπορεί να έχουν αντιδράσεις ή ενστάσεις ε, για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε σχέση με κάθε ένα εθνικό πολιτικό αρμόδιο όταν ακούνε καθημερινά από αυτόν ότι όλα τα αρνητικά προέρχονται από την Ευρώπη και ότι όλα τα καλά λέει είναι του κράτους τους που παράγονται και δημιουργούνται στο ίδιο το κράτος. Ε πώς μπορεί έτσι λοιπόν να υπάρξει δυνατότητα ε, καταπολέμησης ε, της ε, κρίσης και μάλιστα από τα ίδια τα κράτη-μέλη αμφιβάλλω αν κάτι τέτοιο θα μπορέσει να είναι το επίπεδο λήψης αποφάσεων εκεί όπου θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να δώσουμε συνέχεια στις προσπάθειές μας. Και αν θέλουμε να είμαστε θετικοί και συμφωνώ με το γεγονός ότι η ανάλυση των όσων περάσαμε έχει πολλά αρνητικά στοιχεία και συμφωνώ για το ότι οι απαντήσεις πρέπει να έχουν θετικά στοιχεία για τη λύση που θα δώσουμε. Αν θέλουμε να είμαστε θετικοί πρέπει να υπάρχει η ικανότητα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που θα αναζητηθεί και θα προαχθεί για να ακολουθηθεί μια διαφορετική οδός και πορεία για την ανάπτυξη ώστε να μην επαναληφθεί μια τέτοια κρίση στο μέλλον όπως αυτή που σημειώθηκε στο παρελθόν. Και ζώντας αυτά τα οποία έχουμε ζήσει. Είμαι ένας από εκείνους που δεν είμαι υπέρ κατά κανόνα του να αυξηθούν τα δικά μας ωφέλη και προνόμια, διότι πιστεύω ότι δεν είναι η χρονική στιγμή και συγκυρία να κάνουμε κάτι τέτοιο και δεν είναι επιπλέον και αναγκαίο αυτό, διότι επακούμεθα σε αυτά τα οποία έχουμε εγώ, επακούμε στα όσα έχω. Όμως να ζητηθεί η Ευρώπη να υπαρκεστεί στο τίποτα και να ζήσει με το τίποτα δεν μπορεί να το κάνει κανείς αυτό. Δεν είναι για μας, για την αύξηση του επιδόματος ή του ε, ποσού για την γραμματεία, γραμματιακή ε, σύνδρομη. Αυτά τα πράγματα <clears throat> δεν μπορεί να τα δεχτούν οι Ευρωπαίοι. Αλλά είμαι κάθετα αντίθετο σου να συρρυκνωθεί, να μειωθεί ο ευρωπαϊκό προπολογισμό. Διότι δεν επαρκεί. Είμαστε υπεύθυνοι του ενό τεσσαρακοστού τη δημόσια δαπάνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσο πιο πειθαρχημένοι και υποπνεύμα μπορούμε να ε, γίνουμε. Πρέπει να μειωθεί ακόμα περαιτέρω αυτό να γίνει ένα κλάσμα του ενός τεσσαρακοστού. Έχουμε ένα προϋπολογισμό που είναι μικρότερο από το ίμιση του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της Γερμανίας. Με ένα τέτοιο προϋπολογισμό δεν μπορεί να λέει κανείς ότι η λιτότητα πρέπει να ε, λειτουργήσει εδώ. Πρέπει η ε, πειθαρχία και η λιτότητα να μπορεί να λειτουργήσει εκεί όπου υπάρχουν περιθώρια. Εδώ η Ευρώπη δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει τις πολιτικές της. Πώς είναι δυνατόν τις μελλοντικές πολιτικές της να μπορέσει να τις χρηματοδοτήσει δεν στείλουμε ένα θετικό μήνυμα στους πολίτες μας και να τους επεξηγήσουμε με αυτό το μήνυμα ότι είναι στην Ευρώπη που χρειάζονται περισσότερα κονδύλια δημοσιονομικά, Μεγαλύτερος προϋπολογισμός και ταυτόχρονα μπορούν να μειωθούν στους εθνικούς προϋπολογισμούς εκείνα τα κονδύλια που δεν χρειάζονται περαιτέρω για μαζικέ αμυντικές δαπάνες και τα συναφή. Όπου πραγματικά τίθεται το ερώτημα σε τι χρησιμοποιούνται και σε τι ωφελούν όλα αυτά και πρεσβείες κρατών μελών σε όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Ποιο είναι το όφελος. Το πιο γελίο, παράλογο πράγμα που είδαμε και να υφίσταται μέσα σε αυτή την χρονική συγκυρία. Περιθώρια λοιπόν για λιτότητα πρέπει εκεί να αναζητηθούν όχι να ψάχνουμε να βρούμε τίτλο που να δικαιολογεί την ύπαρξη κάποιου διπλωμάτη και το έργο του ενώ δεν υπάρχει. Υπάρχει περιθώριο εδώ και που μπορεί πραγματικά να πιστούν οι Ευρωπαίοι γιατί πρέπει να αυξηθεί ο ευρωπαϊκό προπολογισμό και γιατί πρέπει να συρρυκνωθούν οι εθνικοί προπολογισμοί διότι έχουν ξεπεράσει πλέον τα όρια του. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε αυτήν την έκθεση. Ευχαριστώ Πρόεδρο Πρωτού δώσω τον λόγο στον Αντολίν. Επιτρέψτε μου σύντομα να αντιδράσω στα όσα είπατε. Επειδή θέλω να διασφαλίσω ότι αυτά τα οποία επεξήγησε ο Όλε Σμιτ εδώ δεν θα παρερμηνευθούν. Πρώτον, νομίζω ότι εμείς οι φιλελεύθεροι απόλυτα συμφωνούμε με τα όσα ακούστηκαν. Είμαστε εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και αν δεν λάβουμε τώρα μέτρα, δεν, δεν ακολουθήσουμε τη σωστή πορεία για το μέλλον, τότε θα υπάρχει ο κίνδυνος που θα ελοχεύει να μην μπορέσουμε ούτε καν να κρατήσουμε αυτό το status quo. Δεν θα μπορέσουμε ούτε καμία πρόοδο να, συνεχί, να ακολουθήσουμε και θα ε, οπισθοδρομήσουμε. Αυτό είναι το σταυροδρόμι στο οποίο βρισκόμαστε. Γι' αυτό θέλουμε να εμβαθύνουμε την ε, συνεργασία και την ολοκλήρωση σε πολλούς τομείς, ε, στα κοινωνικά, στα δημοσιονομικά, τα οικονομικά, Τούτων λεχθέντων φυσικά θέλουμε να το κάνουμε αυτό με έναν τρόπο που θα είναι εφικτό να περάσει ως μήνυμα σαν μια επιτυχής αναγκαία βέβαια πρωτοβουλία αλλά και επιτυχής πρωτοβουλία προς τους πολίτες. Πρέπει να διασφαλίσουμε λοιπόν εμείς ότι εμείς θα είμαστε εκείνοι που θα τους πάρουν οι πολίτες στα σοβαρά, εμάς και τις δράσεις μας. Και αυτό απαιτεί αυτό που είπατε, να άρουμε τις αναποτελεσματικές μεθόδους και το κόστος που προκαλείται από τη γραφειοκρατική επιβάρυνση. Πράγμα που δεν είναι καθόλου αναγκαίο να υπάρχει αυτή η επιβάρυνση. Και σε σχέση με μερικά χρόνια πριν, όταν στραφήκαμε στο να δούμε πώς ε, διαθέταμε τα μέσα και τα κονδύλια σε αυτό το σώμα πρέπει να πω ότι πόρο απέχουμε από την ε, βέλτιστη χρήση. Συμφωνώ μαζί σας, δεν πρέπει να έχουμε μεγαλύτερο επίδομα γραμματείας και γι' αυτό στο Κοινοβούλιο επιστρέφω κάθε χρόνο 35% αυτών των επιδομάτων των ενισχύσεων διότι δεν, τις χρειάζομαι, δεν τα χρειάζομαι αυτά τα ποσά και αυτό είναι αυτό το οποίο λέμε εμείς και γι' αυτό το διατυπώσαμε με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να διασφαλίσουμε επαρκή χρηματοδότηση από του ίδιου πόρου. Είτε αυτό θα είναι 3% είτε οποιοδήποτε ποσοστό. Πρέπει να το βρούμε και αυτό να θεσπίσουμε. Αλλά δεν μπορούμε και τουλάχιστον θα είναι δύσκολο να το πούμε στου πολίτε μα, ότι 5 ή 10% να είναι και να συνεχίσουμε να δρούμε με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να το επεξηγήσω αυτό. Δεν είναι ότι δεν βλέπουμε την ανάγκη η Ευρώπη να ακολουθήσει σε νέα βάθρα μια νέα πορεία. Είναι σαφέ αυτό. Θέλουμε να γίνει αυτό. Αλλά όταν έχουμε το θέμα των φόρων. Δεν είμαστε υπέρ του εναρμονισμού των φόρων ή των ποσοστών. Είμαστε υπέρ της ανάπτυξης ενός κοινού βασικού πλαισίου ως φορολογικής βάσης. Μετά ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών ας διαμορφώσει ένα πλαίσιο, κάθε κράτος να θεσπίσει ένα δικό του ποσοστό για τον φόρο αυτό, τη φορολογία αυτή από πλευρά του. Έναν ανταγωνισμό ευδιάκριτο και θα έλεγα καθαρό, να μπορεί να συγκρίνει κανείς συγκρίσιμα πράγματα και όχι μη συγκρίσιμα. Αν πάρει κανείς το 12,5% του Ιρλανδικού φόρου, αυτό μπορεί ουσιαστικά να είναι υψηλότερο ποσοστό από ό,τι σε άλλα κράτη-μέλη, διότι η φορολογική βάση είναι διαφορετική. Λοιπόν, τούτον λεχθέντον δεν θέλω να εξετάσω όλα τα σημεία συνολικά. Αλλά για να διασφαλίσω ότι δεν θα υπάρξει το λανθασμένο μήνυμα που θα περάσει, τα λέω αυτά. Είμαστε υπέρ της προάσπισης της βασικής γραμμής που εκθέτει και παρουσιάζει η Περβάνς. Να έχουμε ένα όραμα για τις ιδέες, για την παρουσίαση των ιδεών μας, πώς πρέπει να μετεξελιχθεί η Ευρώπη στο μέλλον. Δεν θέλουμε δηλαδή να συνεχιστούν τα πράγματα ως έχουν ή να συνεχιστεί το παιχνίδι έτσι. Ο Αντολίν, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω ε, ζητώντας, ε, συγχαίροντας την Περβάνς για την εξαιρετική έκθεση που μας παρουσίασε. Και επίση να περάσω σε αυτή τη συζήτηση για το αν η απάντηση είναι περισσότερη Ευρώπη. Νομίζω ναι, περισσότερη Ευρώπη. Και διαφέρω από τον ε, Όλε Σμιτ. Περισσότερη Ευρώπη για όλα όσα συμβαίνουν. Και γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει η Ευρώπη. Και η Ευρώπη δεν είναι το Ευρωπαϊκό ευρωπαϊκό σύστημα δεν είναι μόνο το κεντρικό ευρωπαϊκό σύστημα. Η Ευρώπη είναι η ενίσχυση των οικογενειών, η ενίσχυση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η ενίσχυση των περιφερειών, των κρατών και φυσικά και της ευρωπαϊκής κεντρικής δομής. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν το ελάχιστο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ελαχιστοποιημένη θέση. Ούτε εγώ βρίσκομαι στην ακραία θέση της μεγιστοποίησης. Θέλουμε τη βέλτιστη πορεία, τη μεσαία βέλτιστη πορεία. Αλλά πόρο απέχουμε από αυτήν σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κοστίζει το ίμιση οποιασδήποτε, ας το πω έτσι, ε, ε, παρουσίασής της. Και γι' αυτό καταλήγουμε στις ε, ε, εφημερίδες και στην ε, πώλησή τους που στοιχίζουν πολλές φορές το διπλάσιο και βρισκόμαστε σε μια πολύ ευάλωτη κατάσταση. Μια κατάσταση πραγματικά μεγάλης οικονομικής αναποτελεσματικότητας που επιβαρύνει τους πολίτες μας, τα συμφέροντά μας, τις αξίες μας και τις αρχές μας και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να επιληθεί και η έκθεση αυτή βρίσκεται σε σωστά ίχνη, σωστή κατεύθυνση. Έχω εργαστεί σε δύο άξονες. Ο ένας αφορά το κρατικό χρέος ο ένας άξονας. Πρέπει να υπάρξει σωστή αναλογία σε σχέση με το κρατικό χρέος, την κρατική υπερχρέωση και το πρόβλημα του οικονομικού τομέα βέβαια από την άλλη πλευρά. Είναι δύο θέματα αλληλοσυνδεόμενα. Πρέπει να ξέρουμε ότι είναι οι δύο του ιδίου νομίσματος και θα ήταν μεγάλος κίνδυνος να δώσουμε προτεραιότητα στην ε, ανάκαμψη του οικονομικού συστήματος με την ενίσχυση του δημόσιου χρέους. Δεν μπορούμε σε σχέση με τα κράτη-μέλη εκείνα να είναι που θα πληρώσουν τα σπασμένα και όλους, ε, όλο το κόστος, διότι αυτό υπονομεύει την αξιοπιστία. Πρέπει να αναζητήσουμε μια σωστή ισορροπία των πραγμάτων. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να καταλήξουμε. Έχουν συστημική σπουδαιότητα τα κράτη. Τα κράτη έχουν θεμελιώδη σημασία στην ευρωπαϊκή δομή και φιλοσοφία και η ανάπτυξή τους με τον ίδιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Με την ίδια ευθύνη και υπευθυνότητα διασφάλισης ενός οικονομικού συστήματος με θετικές συνθήκες και όρους και προϋποθέσεις για να μπορεί να ανταποκριθεί στο παιχνίδι και στις προκλήσεις με αυτή την κατεύθυνση πρέπει να προχωρήσουμε στην ανικοδόμηση του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Και σε σχέση με τα όσα προτείνεται για το, ευρωπαϊκό νομισματικό, για το παγκόσμιο νομισματικό σύστημα, η ρήξη του συστήματο του Bretton Woods όσον αφορά το νομισματικό οικονομικό ε, πεδίο ε, με, τρία, επιτόκια, με το αποθεματικό, με το, τις ε, ε, ισοτιμίες των νομισμάτων, νομίζω αυτά είναι τα κυριότερα σημεία. Και να πούμε ότι υπάρχει ένα τελευταίο τμήμα για τα φορολογικά θέματα όπου έγινε λόγος ότι πρέπει να είναι συγκρίσιμα είπατε. Πρέπει να είναι συγκρίσιμα αλλά επίσης πρέπει να αποφύγουμε κάτι το σκανδαλώδες δηλαδή ακραίες θέσεις για να μπορέσουμε να πετύχουμε ε, τους κοινούς μας στόχους. Προφανές αυτό και πρέπει να καταλήξουμε πέρα από την οικονομική διακυβέρνηση σε μια Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Εκεί πρέπει να δούμε περισσότερα τι μπορούν να γίνουν. Η πρόταση Μόντι είναι αναγκαία συνθήκη αλλά όχι επαρκής και πρέπει να πάμε πιο πέρα. Η Ευρώπη επίσης πρέπει να προτείνει στους πολίτες της κάτι παραπέρα από μια ενιαία εσωτερική αγορά. Οι πολίτες χρειάζονται την οικονομία για να ζήσουν, αλλά δεν ζουν αποκλειστικά μόνο από την οικονομία. Η Ευρώπη είναι κάτι παραπάνω από μια οικονομία. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα new deal, μια νέα οικονομική συμφωνία. Τώρα είναι η χρονική στιγμή για να το κάνουμε αυτό. Η χρονική στιγμή για την ανάπτυξη τη απασχόληση. Μια διαφορετική Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με εκείνη που είχαμε για την οικονομική ανάπτυξη μέχρι σήμερα. Ένα νέο οικονομικό πρότυπο. Να εργαστούμε για όλα αυτά. Αλλά τίποτα από αυτά Τίποτα από αυτά δεν θα είναι εφικτό αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η Ευρώπη ήταν εφικτή επειδή υπήρξε μια μεγάλη κοινωνική συμφωνία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Συμφωνήθηκε αυτό το, αυτή η οικονομική συμφωνία. Ποια θα είναι η παραγωγικότητα, ποια θα είναι τα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών, πώ θα επιμεριστούν τα βάρη σε σχέση με του πολίτε, φορολογικά βάρη παράδειγμα, και ποιο θα είναι το σύστημα ευημερία, το κοινωνική ευημερία που θα ισχύει. Αυτό ήταν το σύμφωνο το οποίο προστα προτάθηκε στους Ευρωπαίους μετά το Δεύτερο Πόλεμο. Μία λύση με απασχόληση, μία λύση με κοινωνική δικαιοσύνη, μία λύση με ένα κράτος ε, ευημερία και εδώ ήταν διαφορετική η Ευρώπη. Αυτές τι απαντήσεις πρέπει να αναζητήσουμε με μια νέα τέτοια συμφωνία τώρα. Ευχαριστώ. Ε, Dank. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ. Κοιτάζω γύρω μου και δεν βλέπω να υπάρχουν άλλοι που να έχουν ζητήσει τον λόγο. Δίνω τον λόγο και πάλι στην Περβάνση παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κάτι μου λέει ότι μάλλον ε, εξακολουθώ και βρίσκονται είναι υπερβολικά πολλέ οι τροπολογίε, ε, αλλά οι πραγματικές συνθήκε τέλο πάντων ίσω να είναι σχετικά πιο άνετε. Και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί φαίνεται ότι για άλλη μια φορά στην Επιτροπή αυτή ο καθένα έχει συνείδηση του μηνύματο που θέλουμε να μεταδώσουμε ενώπιον της ανησυχίας που διαβλέπουμε πάρα πολλούς από τους συμπολίτε μας, υπάρχουν δύο ε, δυνατές προσεγγίσεις. Μία προσέγγιση που οδηγεί ε, στο λαϊκισμό, μια ψήφο που οι δημοκράτες δεν μπορούν να, χαίρονται που βλέπουμε να εξαπλώνονται σε πολλά κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του δικού, της δικής μου χώρας και μια προσέγγιση που στο ότι, που βασίζεται στο ότι ενώπιον μια τέτοια δυσκολία θα πρέπει να διπλωθούμε. Η θέση τη Επιτροπή αυτή είναι ακριβώ να αποδείξει ότι και έχει όραμα, αλλά και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Ότι ενώπιον της πολύ μεγάλη κρίση που βρισκόμαστε, το χειρότερο θα ήταν να διπλωθούμε στο εσωτερικό μας Ενώπιον λοιπόν αυτή τη κρίση, που είναι η πρώτη μεγάλη κρίση μετά την παγκοσμιοποίηση, κατά τη διάρκεια τη παγκοσμιοποίηση, θα πρέπει πλέον να, λάβουμε υπόψη ακριβώ αυτό το παγκόσμιο επίπεδο τη κρίση την οποία βιώνουμε. Ευχαριστώ το σύνολο των συναδέλφων για όσα είπαν και κρατώ από την ε, παρέμβαση εξ του ΕΛΚ, του κ. Καράς, σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα συμπεράσματα της ε, Επιτροπής ε, σε ό,τι αφορά θέματα του προπολογισμού. Στο θέμα του προπολογισμού του Ευρωπαϊκού είναι διαφορετικέ προσεγγίσεις. Τι θα κάνουμε εν τη επόμενη χρήση και τι μπορούμε να προτείνουμε σε πιο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Πάντως το μοντέλο σε ό,τι αφορά τους ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να δεσμευόμαστε αν θέλετε, με την παράλληλη αυτή προσέγγιση, νομίζω είναι κάτι που πρέπει να το μελετήσουμε εκ του σύνεγγης. Σε ό,τι αφορά την σημασία της θεματικής περί ενέργειας και περιβάλλοντος, σε σχέση με την ε, παρέμβαση Κομφαράτη, δεν μπορώ να υποστηρίξω τις θέσεις. Το είπατε κι εσείς, κύριε Πρόεδρε, και θα επανέλθω σε αυτό, πάνω σε δύο-τρία θέματα. Ο Φρανκ Έγγελ επανέλαβε, ξαναπήρε αν θέλετε την μπάλα σχετικά και ε, αντέδρασε στην εισήγηση Σμιτ, σύμφωνα με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι απάντηση σε όλα. Πιστεύω πραγματικά ότι σίγουρα δεν είναι αυτό το οποίο ευχόμαστε. Εάν ε, ήθελα να αναπτύξω περισσότερο και πιο αρθρωμένα μια απάντηση απέναντι σε αυτήν την ανησυχία, θα έλεγα ότι αυτή του είδους, αν θέλετε, η διακυβέρνηση είναι, θα έλεγα, πολύ επίπεδη. Αυτός είναι ο κατάλληλος όρος. Και υπάρχει μια πραγματική δυσκολία, την οποία, αν θέλετε, μπορούμε επαρκώς να αντιμετωπίσουμε και να τη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά όταν λέει ο πρόεδρος Μπαρόζο ότι για να καλύψουμε το κενό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υπάρχει κινητοποίηση διαφόρων φορέων σε διάφορα επίπεδα, ακριβώς αυτό είναι, ότι πρέπει να φρώσουμε καλύτερα σε ό,τι αφορά τη συνέχεια και τη συνέπεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι πολλές λύσει λύσεις σε αυτή την κρίση θα εξαρτηθούν ε, παραδείγματι από την κινητοποίηση τοπικών αρχών. Το είδαμε σε απαντήσεις στην κρίση, άμεσες ε, απαντήσεις σε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό. Πολύ συχνά είναι οι τοπικές κοινότητες, αυτές που είναι αν θέλετε στη βάση, που μπόρεσαν να κινητοποιήσουν τις απαραίτητε ενέργειες και δράσεις για να υπάρξουν απαντήσεις και προφανώς βέβαια μακριά από εμά η όλη ιδέα του να εμποδίσουμε κάτι τέτοιο στο μέλλον. Το αντίθετο. Σε ό,τι αφορά τον όμιλο των 20, τον G20, ε, και εγώ θέλω, θα πρόκειται να, να, οργανωθεί μια ειδική συνάντηση ε, εν ώψη τη στρατηγική που θα πρέπει να εκπονηθεί. Θα πρέπει να κρατήσουμε ακριβώς την ιδέα του να υπάρχει μια πολύ καλύτερη παγκόσμια διακυβέρνηση δεν αποδέχομαι το επιχείρημα το οποίο ανέπτυξε ο συνάδελφος Σβίμπερν που είπε ότι θα είναι δύσκολο να ζητήσουμε πράγματα από την Αμερική και τη, από τους Αμερικανούς και τους Κινέζους και πρέπει να κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Μα όχι αγαπητή συνάδελφοι, δεν μπορούμε να αφήσουμε τους Αμερικανούς και τους Κινέζους να συνδιαλέγονται μεταξύ τους και εμείς να είμαστε αν θέλετε ή ο, ο αμέτωχος, ε, ο απέξω ο καθώς παρακολουθεί ή να μην ή να υφιστάμεθα όσα έχουν αποφασίσει. Έχουν τελείω διαφορετική φάση και προσέγγιση ό,τι αφορά την παγκόσμια αγορά και πρέπει και εμεί να βγούμε σε αυτή τη μάχη. Και για να έχουμε διαπραγματευτική ισχύ για να συζητήσουμε μαζί του και για να έχουμε σαν στόχο ακριβώ να μπορούμε να, να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι. Σε σχέση με αυτό λοιπόν, ο όμιλο των 20 είναι κρίσιμο ζήτημα. Γιατί όπω το γνωρίζετε, ορισμένε φορέ αν θέλετε, είμαστε και συγχρονόμονες από αυτού και εγώ είμαι. Θεωρώ ότι ο όμιλο των 20, το G20 είναι ένας χρήσιμο μηχανισμός, ένα χρήσιμο εργαλείο ως ε, ένα χώρος, αν θέλετε, ένα φόρο που γίνεται ανεκτό στα πλαίσια παγκόσμια κυβέρνηση από την Κίνα αλλά δεν είναι ικανοποιητικό θεσμό για την ανάπτυξη αυτή τη παγκόσμια διακυβέρνηση. Δεν μα δίνει τα απαραίτητα εργαλεία και παραμένει, και παραμένει να έχει μια ατζέντα διακυβερνητική, πω εκ τούτου δεν μπορεί να συμπεριλάβει το σύνολο των προβληματικών του πλανήτη. Εξού και η όλη ιδέα να υπάρξει μια, ένας μετασχηματισμός, αν θέλετε, αυτού του ομίλου. Οι Ευρωπαίοι ίσως ε, να ζητούν ακριβώς τη συγκεκριμένη θέση πέντε αν θέλετε στις 20 θέσεις να μπορούν να δώσουν, να δώσουν αν θέλετε στα σπάργανα ένα είδος θεσμού αν θέλετε που θα αφορά την οικονομική διακυβέρνηση στα πλαίσια της ε, πλανητικής αν θέλετε αυτής διακυβέρνησης. Στα σχέση με τη, τα, τα προωθούμενα από τον Μάριο Μόντι που αναφέρθηκε προηγουμένως σέβομαι απόλυτα και το γνωρίζετε, ξέρετε πολύ καλά την εκτίμηση και σεβασμό που έχω απέναντι στον Επίτροπο. Θεωρώ όμως ότι σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, το ευρωπαϊκό σχέδιο, το ζήτημα της εσωτερικής αγοράς δεν είναι επαρκές για να οργανώσουμε τις προβλέψεις και το όραμά μας. Αυτό που είχαμε πει στην, ε, στην πρώτη έκθεση που συντάχθηκε σχέση με την κρίση είναι προ αυτή την κατεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα απαραίτητο κατόφλι, αν θέλετε, απαραίτητη πλατφόρμα για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά σχέση με τι μολυντικέ προκλήσει, το ζήτημα του πώς θα μπορέσουμε ακριβώς να χρησιμοποιήσουμε την ευρωπαϊκή εικονότητα για να προχωρήσουμε στην παιδεία, στην έρευνα, στην καινοτομία, στις υποδομές, στην ε, ανεξαρτησία στον ενεργειακό τομέα, την συνεισφορά μα στην ε, αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού ζητήματο, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αμυγό σαν ένα ζήτημα απλώ εσωτερικής, ενιαία εσωτερική αγορά. Αυτό είπαμε εξ αρχής και πρέπει να παραμείνουμε σε αυτό το πνεύμα. Κατά τον ίδιο τρόπο, σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ σα παραπέμπω και σε παρατήρηση του συναδέλφου Όλε Σμιτ, σε επίπεδο ενωσιακού προπολογισμού. Κανείς δεν μπορεί, δεν προτείνει έτσι αφηρημένα από ένα αφηρημένο φεντεραλιστικό όραμα που θα ήταν που θα ήταν άσχετο με την όλη πραγματικότητα να μιλήσουμε για διαφορετικό προπολογισμό. Γιατί τα συμπεράσματα που είχαμε υιοθετήσει στην πρώτη έκθεση, αυτό το οποίο λέγαμε ακριβώ, είναι ότι εκεί που υπάρχουν μοιρασμένε αρμοδιότητε θα πρέπει να είναι εργό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν έχουμε συμφωνήσει σε αυτό, πρέπει λοιπόν να υποστούμε και τι ανάλογε συνέπειε. Ο προπολογισμό που έχουμε σήμερα δεν είναι επαρκή για κάτι τέτοιο. Βέβαια, αυτό σημαίνει, αν θέλετε, μεγαλύτερη ισχύ. Κάποια μέρα, ξέρετε, εγώ δεν θα είχα ποτέ εμπιστοσύνη στον πρόεδρο Μπαρόζο για να διαχειρίζεται ένα προπολογισμό, αν θέλετε, που θα είναι 100% του ΑΕΠ, κάθε άλλο. Αλλά πάντω ο στόχο προ εκεί ε, κατευθύνεται, ανάλογα με τι αρμοδιότητε που θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σχέση με τις προτάσεις ε, του συναδέλφου, σκεπτόμενοι τις ε, λειτουργίες και τις αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σε πολλούς πολίτες της μέρες μας μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να φαίνεται περισσότερο πρόβλημα παρά λύση, εν αναμονή, εν πάση περιπτώσει, εγώ θα εξακολουθώ να υποστηρίζω και να, φω, και να ζητώ κάθε, κάθε μία από τις χώρες μας, ναι, να είναι η χώρα μας εθνική, αλλά η Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη είναι το μέλλον μας. Χαίρομαι, λοιπόν να προτείνω σε όλους τους σκιώδεις ε, εισηγητές και εισηγητές γνωμοδότησης να προτείνουμε ένα χρονοδιάγραμμα ώστε να έχουμε ε, το βέλτιστο και καλύτερο δυνατό σχετική ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για τους δύο συναδέλφους που ήρθαν τώρα στο τέλος πρέπει να πω δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Ήταν μια σύντομη αλλά πολύ παραγωγική συνεδρίαση αυτή είχαμε σκεφτεί αν θα έπρεπε να διατηρήσουμε τη σημερινή ημερομηνία ή θα αποσύραμε τη συνεδρίαση αυτή την ακυρώναμε. Ήταν πολύ χρήσιμη, πραγματικά γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και είχαμε και νέες σκέψεις που ακούσαμε και παρουσιάστηκαν. Και χαίρομαι και προσβλέπω στην αντιμετώπιση και εξέταση των τροπολογιών. Και είμαι σίγουρος ότι αυτή τη φορά σχετικά σύντομα, σχετικά γοργά θα έχουμε ικανοποιητική συμφωνία στην οποία θα καταλήξουμε. Μέχρι αύριο λοιπόν τροπολογίες. Επόμενη συνεδρίαση 5 Μαΐου και μετά 23 Μαΐου. Και αρχές Ιουνίου νομίζω θα ψηφίσουμε. 30 Μαΐου θα ψηφίσουμε. Εντάξει. Σας ευχαριστώ. Καλή μέρα. Γεια σας.